Ευχαριστώ. Κύριο Κού, ένα λεπτό. Παρακαλώ κύριε Κού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όταν πριν από 14 χρόνια γίνατε υπουργό οικογενειακών υποθέσεων, η γυναίκα μου και εγώ χαρήκαμε πολύ γιατί ξέρουμε ότι έχετε 7 παιδιά και εμείς τότε περιμέναμε το δέκατο μας παιδί και περιμέναμε ότι θα βοηθούσατε τις οικογένειες αλλά δυστυχώς απογοητευθήκαμε ικτρά και όταν ε, άκουσα σήμερα την ομιλία σας ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια Ευρώπη με βάση την ελληνική φιλοσοφία και το ρωμαϊκό δίκαιο αλλά κάτι λείπει, ε. Δεν άκουσα τις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης να αναφέρεται. Χωρίς αυτές δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θα καταρρεύσει. Αυτό το οικοδόμα θα γίνει νέος πύργος της Βαβέλ. Ή ένα οικοδόμημα που θα καταρρεύσει όπως είπα. Γιατί έχει σαθρά θεμέλια. Θα πρέπει να αποφευχθεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει μια ταπεινωτική διαδικασία δυνάμη του άρθρου 7 κατά της Πολωνίας. Κάποιος αποφάσισε ότι είναι νομότυπο όταν, για παράδειγμα, οι δικαστές δέχονται την απαλωτρίωση περιουσία, την κλοπή περιουσίας ε, ε, ηλικιωμένων ανθρώπων. Και από την άλλη πλευρά είναι παράνομο όταν κάποιοι επηρεάζουν το δικαιικό σύστημα. Για παράδειγμα, ε, ε, γίνεται τυχαία η κατανομή των υποθέσεων στο δικαστήριο και κάθε φορά που ρωτάω, δείξτε μου, δείξτε μου έστω και ένα παράδειγμα. Ένα, όχι οχτώ, όχι δέκα παραδείγματα. Ένα και μόνο παράδειγμα της λύσης που εμείς εφαρμόσαμε στην Πολωνία που, και που δεν υπάρχει ήδη και δεν εφαρμόζεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και πάντα λαμβάνω την ίδια απάντηση. Σιωπή. Σιωπή. Γι' αυτό και σας ρωτάω κύριε Υπουργέ, εσείς θα τερματίσετε αυτή την γελία πολιτική δράση του άρθρου 7. Σας ευχαριστώ κυρία Σούιτσα, Ντούμπραφκα Σούιτσα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φοντερ Λάιεν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγική σας ομιλία και θα ήθελα και πάλι να σας υπενθυμίσω ότι ίσχυε η διαδικασία Σφίτσεν Τι Είχαμε το δικό μας κορυφαίο υποψήφιο, τον κύριο Μάνφρετ Βέμπερ. Και δυστυχώς αυτοί που ε, κάνουν τους μεγάλους δημοκράτες δεν την δέχτηκαν αυτή τη διαδικασία και διόρισαν εσάς. Και όμως ε, είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστή η διαδικασία του, του and Ε, και χαίρομαι που μας είπατε ότι εσείς θα σεβαστείτε στο μέλλον αυτή την ε, αρχή του Speech Candidate. Χαίρομαι που είστε γυναίκα, ε, χαίρομαι που δώσατε έμφαση στην ισότητα των φύλων, μιλήσατε για τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι θα προωθήσετε τα δικαιώματα του μισού πληθυσμού της γης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι γυναίκες ελπίζω στο μέλλον να μιλήσετε περισσότερο και για κάτι που θα πω τώρα. Ε, είμαι Κροάτισσα. Ε, μιλήσατε για την ε, ανάγκη ενότητας, αλλά δεν ε, μιλήσατε για τις διαφορές μεταξύ ε, Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου, Ευρωζώνης και μη Ευρωζώνης, χώρου Σέγγεν και χωρών εκτός του χώρου Σέγγεν. Ελπίζω να επενδύσετε χρόνο και ενέργεια για να διορθούν και αυτές οι διαφορές. Επίσης, για τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια, την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ε, είπατε επίσης ότι η οικονομία θα πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι την οικονομία. Χαίρομαι γι' αυτό που είπατε. Και επίσης ε, δεν μπορούμε να ξοδεύουμε περισσότερα από αυτά που έχουμε κερδίσει. Πρώτα θα πρέπει να βγάζουμε χρήματα και μετά να τα ε, δαπανούμε και να τα κατανέμουμε. Χαίρομαι για όλα αυτά. Επίση, χαιρόμαστε και για τον Green Deal που προτείνατε, αυτή την οικολογική συμφωνία. Παρόλο που οι πράσινοι δεν θα σα υπερψηφίσουν. Το Green Deal είναι σημαντικό για τι επερχόμενε γενιέ, για τα παιδιά μα. Και χαίρομαι που θα είναι και αυτό το τμήμα του χαρτοφυλακίου σα. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, θα προτιμούσα να συνεχίσετε το σχέδιο για την Αφρική ο κύριος Βέμπερ μάλιστα στο προεκλογικό του πρόγραμμα είχε ειδικό επίτροπο για την Αφρική. Μακάρι να το αισθενιστείτε κι εσείς αυτό. Γιατί θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτή τη σημαντική ήπειρο και για την Ευρώπη. Εμείς θα σας υπερψηφίσουμε, θα σας στηρίξουμε και επίσης ε, θα, θα πρέπει ε, να θυμόμαστε αυτό που μας ενώνει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευχαριστώ. Ειρήνη και ευημερία. Σε ο, ε, ο κύριος Μορένο Σάντσες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύρια Φόντερ Λάιεν, καλωσορίσατε στο οίκο στον οίκο των Ευρωπαίων πολιτών, ανδρών και γυναικών. Εσείς δεν ήσασταν καντιντάτ, ούτε είστε σοσιαλίστρια προς το παρόν. Μετά στο τέλος της θητείας θα δούμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, γνωρίζετε ότι η πρόσβαση στη θέση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περνάει από το σοσιαλιστικό δρόμο. Και από ό,τι φαίνεται ότι εσείς είστε διατεθειμένοι να συμβαδίσετε μαζί μας ε, με τις δεσμεύσεις που εχθές εξέδωσε η ομάδα μας και που ε, αναλάβατε και εσείς σήμερα το πρωί εδώ στην Ολομέλεια. Η θητεία σας λοιπόν θα έχει σοσιαλιστικό αποτύπωμα με μεγαλύτερη ε, κοινωνική δικαιοσύνη, με κατώτατο ευρωπαϊκό μισθό, με ε, ασφάλεια για την ε, ε, ευρωπαϊκή ανεργία και μια εγγύηση για τους νέους και για τα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζουμε επίσης τη στρατηγική σας για την ισότητα των φύλων. Με την άρση των μισθοδογικών φραγμών, η μάχη των γυναικών κατά της βίας από τους άνδρες και φυσικά το να προσπαθείτε να έχετε ισότητα των φύλων στο μελλοντικό σώμα των Επιτρόπων. Κυρία Φοντερ Λάιαν, αν εκλεγείτε θα προχωρήσουμε μαζί για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις σας με οδηγίες, με κανονισμούς, με μέσα και τα κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους. Κυρία Φοντερ Λάιεν, εάν λοιπόν εκλεγείτε θα συνεργαστούμε με μεγάλη ευχαρίστηση με την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας ευχόμαστε πολύ καλή τύχη στα γερμανικά. Ευχαριστώ η κυρία Κατάινεν για ένα λεπτό. Ε, σας παρακαλώ να σεβαστείτε όλοι του χρόνου αγόρευσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Βαντερ Λάιεν. Στο πρόγραμμά σας έχετε θέσει ως προτεραιότητα τα κλιματικά θέματα. Και σε αυτή τη συζήτηση εδώ ε, οι συνάδελφοι μας ζητούν συγκεκριμένα μέτρα, δράσης και λύσεις. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα και εγώ να επικεντρωθώ στο κλίμα και κυρίως σε δασικά ζητήματα, διότι ε, είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να έχουμε μια Ευρώπη χωρίς άνθρακα και να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής ενέργειας και κλίματος το όρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2050, τα ε, βιοκαύσιμα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για να σταματήσουμε να εξαρτώμαστε από την ε, οικονομία των ε, ορυκτών καυσίμων. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προστασία λοιπόν και να υπάρχουν και ενεργή και βιώσιμη δασική διαχείριση και όχι μέσω του περιορισμού της χρήσης της ξυλίας. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω πώς θα εξασφαλίσετε εσείς ότι στην Ευρώπη η χρήση ξυλίας ε, θα θεωρείται ως πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τι άποψη έχετε εσείς γι' αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κολάγια για ένα λεπτό. Ο κύριος Κολάγια, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φοντερ στην τελευταία δημόσια διαβούλευση ε, οι ενδιαφερόμενοι και οι πολίτες απέρριψαν ε, το καθεστώς ε, ευθύνης ε, της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όπως θα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, απόδοση ευθυνών για όσους παρέχουν διαδικτυακό περιεχόμενο ήταν ένα από τα επίμαχα ζητήματα ε, στην τελευταία μεταρρύθμιση για τα πνευματικά δικαιώματα. Πάνω από 250.000 άνθρωποι μόνο στη Γερμανία διαμαρτυρήθηκαν κατά του λεγόμενου άρθρου 13, το οποίο είναι τώρα το άρθρο 17 της Οδηγίας για τα Πνευματικά Δικαιώματα και ε, την εισαγωγή συγκεκριμένων φίλτρων. Πάνω από 5 εκατομμύρια υπέγραψαν την αίτηση που είναι η μεγαλύτερη στην ευρωπαϊκή ιστορία. Ε, σε αντίθεση με όλα αυτά, στο πρόγραμμά σας για την Ευρώπη φαίνεται ότι είστε υπέρ ε, της νέας συζήτησης της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και λέτε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσετε τους ε, κανόνες ευθύνης και ασφάλειας. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει αναβάθμιση αυτών των κανόνων και επίσης την αρχή του ασφαλούς λιμένα για παρόχους υπηρεσιών, η οποία λέτε ότι θα μείνει άθικτη και δεν θα υπάρχουν επιπλέον φίλτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μπέκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η Ευρωζώνη μαζί με την Ιαπωνία έχουν το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και τους υψηλότερους φόρους του αναπτυγμένου κόσμου. Ένας φόρος για το διοξείδιο του άνθρακο για την Ένωση απαιτεί ομοφωνία. Κύριε Υπουργέ, εσείς θέλετε να αμφισβητήσετε την αρχή αυτή της ομοφωνίας. Το Υπουργείο σας σπατάλησε δισεκατομμύρια για εξωτερικούς συμβούλους, ιδιαίτερα έναντι, πλήρωσε την εταιρεία συμβούλου McKinsey. Μόνο το 1 τρίτο του εξοπλισμού της, του στρατού της Γερμανίας ε, λειτουργεί. Ε, Κάποιο δημοσιογράφο έγραψε ότι η εταιρεία McKinsey χρησιμοποιεί ε, το γερμανικό στρατό ως ε, μηχάνημα απόσυρση μετρητών. Πληρώνουν οι φορολογούμενοι, καταστρέφεται ο στρατός και τσεπώνει η McKinsey. Μήπως θα έπρεπε να δούμε μέσω κάποιας ε, μελέτης πώς εφαρμόζεται η κλιματική πολιτική και η πολιτική ασύλου ε, στη Γερμανία ε, προς το συμφέρον της Ένωσης. Θα ήθελα να το μάθουν οι πολίτες μας. Βόντρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, στην ομάδα μας σας άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα και θεώρησα ότι υπήρχε ελπίδα αλλά διαβάζοντα τα γράμματά σα χθε και ακούγοντα την ομιλία σα σήμερα, ομολογώ ότι απογοητεύομαι όλο και περισσότερο. Υποχωρήσατε πλήρως έναντι της, ε, του θεματολογίου και των προτεραιοτήτων των ε, πρασίνων και των προοδευτικών. Το 95% των απαιτήσεων των πρασίνων το δεχτήκατε και θέλουν να σε βάλουν το άλλο 5% και από ό,τι φαίνεται θα το κάνετε. Αντί να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή, συμφωνείτε με αυτούς τους ε, ανέφικτους στόχους για το 2030 και λέτε ότι θα πρέπει να έχουμε μια κοινωνία χωρίς εκπομπές άνθρακα. Εγώ είμαι από την Τσεχοσλοβακία. Αυτό μου θυμίζει αυτά που λέγανε παλιά στην ε, Τσεχοσλοβακία για την αταξική κοινωνία. Όλα αυτά είναι αφύσικα. Πριν από 30 χρόνια στην ε, Κίνα όλοι είχαν ποδήλατο ενώ στην Ευρώπη όλοι είχαν αυτοκίνητο. Θεωρείτε το 2030 στην Ευρώπη αυτοκίνητα θα έχουν μόνο δισεκατομμυριούχοι ηλεκτρικά φυσικά, ενώ οι υπόλοιποι θα επανέλθουμε στα ε, ποδήλατα, ενώ στην Κίνα βέβαια όλοι θα έχουν αυτοκίνητα. Αυτό είναι το όραμά σα για την Ευρώπη. Έτσι θα είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη με την Κίνα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σον Κέλλη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φοντελάιν, ελπίζω να τα πάτε καλά. Πριν από δύο εβδομάδες σας άκουσα, αλλά και αυτό που είπατε σήμερα επιβεβαιώνει την άποψή μου ότι ε, είστε καταπληκτικοί. Έχετε μεγάλο ταλέντο, έχετε αυτοπεποίθηση, έχετε όραμα, είστε ήρεμοι, είστε πλήρως εξοπλισμένοι για να επιτελέσετε τα καθήκοντά σας που ελπίζω να ε, σας τα εγκρίνουν τουλάχιστον 400 συνάδελφοι σήμερα το απόγευμα. Αναφέρατε πολλούς τομείς μεγάλης σημασίας. Ο σημαντικότερος, ε, η σημαντικότερη ανησυχία των πολιτών ε, κατά τις εκλογές ήταν η κλιματική αλλαγή και χαίρομαι που θα το αντιμετωπίσετε. Και θέλω να σας ρωτήσω, όσο πηγαίνουμε προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, θα φροντίσετε να μην ξεχάσουμε κανένα, να υπάρξει μια δίκαιη μετάβαση για όλους και οι αγρότες στην Ιταλία και οι ε, ανθρακορίχοι στην Πολωνία και οι δικοί μου συμπολίτε. Αναφέρθηκε το θέμα των Spitzenkandidat, μα εσείς είστε και θύμα και ε, ωφελείστε από αυτό. Μήπως θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια ομάδα εργασίας με εκπροσώπους και από τα τρία θεσμικά όργανα ούτω ώστε να εκπονήσουμε μια καλύτερη λειτουργία του συστήματο αυτού για το μέλλον, ούτω ώστε να διασώσουμε αυτή τη διαδικασία. Επίση, χάρηκα για αυτό που είπατε για τον Brexit και για τη συνέπεια που έχετε επιδείξει στι απαντήσει που δώσατε στην ομάδα μα, στο ΕΛΚ και που αναλαμβάνετε σήμερα για το backstop, για τη συμφωνία αποχώρηση και για την ευελιξία όσον αφορά την ενδεχόμενη παράταση για την αποχώρηση. Θα ήθελα να πείτε περισσότερα για τη στήριξή σας ε, και στο μέλλον για την Ιρλανδία. Γιατί από τον Γιάνν Κλοντ Γιούμπερ και τον Κλοντ Μπαρνιέ είχαμε ε, απαρασάλευτη υποστήριξη. Και επίσης ε, αυτά που είπατε για την ισότητα των φίλων ε, είναι κάτι το οποίο σίγουρα με βρίσκει σύμφωνο και είστε στην κατάλληλη θέση για να τα προωθήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λιμπεράτσκι, Μπογκούσουαφ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φοντερ Λάιεν, ε, ως ε, Πολωνός Σοσιαλδημοκράτης, θα ήθελα να πω ότι με κάθε, φορά, ε, κάθε φορά που ξαναβλεπόμαστε και έχουμε νέα επαφή μαζί σας, αυξάνεται και η συμπάθειά μας απέναντί σας. Πάντως, χωρίς δεσμεύσεις ε, χωρίς ε, δέσμευση υπέρ του κλίματος ε, και χωρίς δέσμευση για το κράτος δικαίου δεν γίνεται. Και χαίρομαι που τα τονίσατε σήμερα όλα αυτά. Και επίσης χαίρομαι που είπατε ότι το κόστος της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να κατανεμηθεί δίκαια. Δεχόμαστε τη θέση σας για, και τις διακηρύξεις σας για την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής και το Ταμείο για, τη δίκαιη, για το δίκαιο μετασχηματισμό. Επίσης, ε, ε, κατώτατος μισθός, να έχουμε παρόμοια κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη. Συμφωνούμε με αυτό. Για την ε, εξωτερική σας πολιτική δεν ακούσαμε την ανατολική διάσταση. Ρωσία, Ουκρανία, τι γίνεται με όλα αυτά. Εκεί έχουμε κάποιο έλλειμμα. Και τέλος, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη γεωγραφική ανισορροπία στην κατανομή ισχύω στα θεσμικά όργανα. Ε, η Γερμανία και η Γαλλία είναι οι πρώτες, μετά στο δεύτερο στρώμα Ολλανδία, Ισπανία, ε, η Πολωνία τίποτα. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε για να διορθώσετε αυτή τη γεωγραφική ανισορροπία να εκλέγετε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκιουτσούκ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φοντερ η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεταρρύθμιση και μετασχηματισμό. Αυτό ήταν το μήνυμα των Ευρωπαίων πολιτών. Απερίφραστο μήνυμα. Είναι σαφές ότι αγαπούν οι Ευρωπαίοι πολίτες την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουν να μεταρρυθμιστεί, να αλλάξει, να γίνει πιο αποτελεσματική και να έρθει πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Οπότε μια καλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα έχει κέρια σημασία. Όχι όμως η ολοκλήρωση αυτή να γίνει εις βάρος της διεύρυνσης. Και σίγουρα η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών Δυτικών Βαλκανίων έχει θεμελιώδη σημασία γιατί είναι μια ε, ζώνη με πολύ ευαίσθητη ασφάλεια. Ε, χωρίς ε, αρμόδιο επίτροπο διεύρυνσης, ε, τι σημαίνει δεν θα έχουμε περαιτέρω διευρύνσεις. Δεν θέλουμε επίσης μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Θέλουμε επίσης μια Ευρώπη με ίδιες προδιαγραφές, όχι διαφορετικά πρότυπα και προδιαγραφές ε, στα τρόφιμα, στις μεταφορές και ούτω καθεξής. Επίσης ε, υπάρχει διαφορά μεταξύ χωρών εντός και εκτός έγκεν. Ε, τι πρόκειται να κάνετε για την κατάσταση αυτή. Η απερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε πολλά, αλλά δεν τήρησε τις υποσχέσεις της. Επίση, θέλουμε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να περάσουμε απρόσκοπτα στο νέο, στη νέα περίοδο προγραμματισμού του 2021. Ο κύριο Κουμπίλιο για δύο λεπτά. Κυρία Φοντελάιν, ε, προέρχομαι από τη μικρή Λιθουανία και ευχαρίστω θα υπερψηφίσω την υποψηφιότητά σα. Ε, γιατί ε, ε, χαίρομαι που μιλήσατε για το ε, ΝΑΤΟ και γιατί έχουμε την παρουσία ε, και γερμανικών στρατευμάτων μέσω του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία για την εξασφάλιση της ασφάλειας. Ελπίζω να, είναι, να είστε συνετοί και αποτελεσματικοί πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε πραγματική ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί για μα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μια κοινή αγορά ε, και δεν είναι μόνο η οικονομική και η κοινωνική μα ευημερία που εξαρτάται από αυτή και τα περιβαλλοντικά μέσα για να καταπολεμήσουμε κλιματικέ αλλαγέ. Τα πλανεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα όταν σε εθνικό επίπεδο αντιμετωπίζουμε όλο και μεγαλύτερες ε, προκλήσεις ε, για μακροπρόθεσμη οικονομική στασιμότητα ε, και εισοδηματικά προβλήματα. Θέλουμε όμως και πολιτική σταθερότητα και έχουμε μοναδικούς μηχανισμούς για να διευρύνουμε το χώρο ασφάλειας, σταθερότητας, κρατούς δικαίου και οικονομικής ευημερίας στην Ευρώπη. Και φυσικά σημαντικό στοιχείο είναι και η διεύρυνση. Εμείς ε, έχουμε με τις επιτυχίες μας δώσει το καλό παράδειγμα για το πόσο ισχυροί είναι οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε ευγνώμονες ε, για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από τη δεκαετία του 90. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας παροτρύνω ε, αν αναλάβετε την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εφαρμόσετε φιλόδοξε πολιτικέ και διεύρυνση προ χώρε των Δυτικών Βαλκαλίων και στη συνέχεια προ χώρε τη Ανατολική Γειτονία, την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία γιατί και οι χώρες αυτές αξίζουν την αλληλεγγύη μας. Και εμείς αξίζουμε ε, ειρηνική και σταθερή γειτονία. Και σίγουρα μια ένα μήνυμα προς την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία για τη διεύρυνση θα είναι ένα μήνυμα για να παροτρύνουμε και τη Ρωσία να κάνει κάποιες θετικές μεταρρυθμίσεις. Και ελπίζω υπό την ηγεσία σας κυρία Φοντερ Λάιν να υλοποιήσετε ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύρια Βαντερ Εκτιμώ ιδιαίτερα την προοδευτική και φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση της σημερινής σας παρέμβασης και την επιστολή που στείλατε στην ομάδα μας. Ως επικεφαλής της ε, Ρουμανικής Αντιπροσωπείας των Σοσιαλδημοκρατών θα σας υπερψηφίσω και να σας πω και γιατί. Για την ελπίδα. Την ελπίδα για τη μάχη κατά των διακρίσεων ε, της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ε, θα πρέπει να δώσετε μια μάχη για να ε, αντιμετωπίσουμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπάρχει ο χώρος Σέγγεν, υπάρχουν πολίτες στην Ευρώπη στα αριστερά και Ρουμάνοι στα δεξιά, οι οποίοι δεν χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων. Ελπίζω λοιπόν να αντιμετωπίσετε αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επίση, ε, πρέπει να ληφθούν και μέτρα στον τομέα τη γεωργία. Γνωρίζετε ότι οι γεωργοί των ανατολικών χωρών έχουν πολύ λιγότερα έσοδα από του ε, υπόλοιπου Ευρωπαίου γεωργού ε, των χωρών τη δύση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πνεύμα ισοτιμίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω να δώσετε κατάλληλου πόρου για τι χώρε οι οποίε βρίσκονται σε διαδικασία ενεργειακή μετάβαση και βιομηχανική μετάβαση. Πρόκειται ε, παιδιά, μητέρες ε, και νέους ανθρώπους οι οποίοι θα πληγούν εάν υπάρξει ενεργειακή ε, ένδυα και δεν υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση. Και αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ κύριο Σπάιτ για ένα λεπτό. Αγαπητή Ούρσουλα Φορνελάιεν, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρότερη ε, και πιο ενωμένη ε, πολιτική εξωτερικής, ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Υπάρχουν πολιτικές οι οποίες γίνονται ασήμαντες ακριβώς λόγω των ελλείψεων στον τομέα αυτό. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δείξει αφοσίωση. Και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει στα ενία της κάποιον ο οποίος έχει εμπειρία στην πολιτική ασφάλεια και άμυνας και θα αντιμετωπίσει και τις ελλείψεις οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν. Ε, όλα αυτά σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ βεβαίως. Η Ούρσολα Φοντερ Λάιεν έχει συμβάλει στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων και στο ανατολικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υποστηρίξω την κυρία Φόντερ σήμερα λόγω της ε, πείρας της σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και γιατί ε, αντιλαμβάνεται και κατανοεί το όραμα ε, μιας ισχυρότερης Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέτσολα για μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το τείχος του Βερολίνου έχει πέσει ε, για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα από όσο ήταν όρθιο. Αυτό βέβαια ε, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν από προσωπικότητες είναι ελπίδα και πέρα από ε, ε, προβλήματα είναι δικαιοσύνη. Είμαστε λοιπόν ισχυρότεροι, είμαστε γενιές ανθρώπων που πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται, αλλά φυσικά πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Δεν είμαστε άμομοι, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει ακόμα να λύσουμε, αλλά είναι πολύ σκληρή η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλούς και πόρο απέχουμε ακόμα από τη λύση. Θέλω η γενιά των παιδιών μου να θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι η λύση, όπω ήταν και για του γονεί μου. Γι' αυτό ακριβώ δεν μπορούμε να σιωπούμε όταν ε, απειλούνται οι θεμελιώδει ελευθερίε μα. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δεχτούμε ότι ε, δημοσιογράφοι όπω η Ντάφνη Καρουάνα Γαλήθια απειλούνται και δολοφοτούνται όπω έγινε πριν από 21 μήνε ακριβώ ε, σήμερα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρείτε ότι είναι αγαθό η δημοσιογραφία. Θα πρέπει οι νέοι άνθρωποι να μην έχουν περισσότερο πλαστικό από ψάρια στη θάλασσέ σου. Πρέπει να βρεθεί μια τολμηρή λύση για το κλίμα και το περιβάλλον σήμερα, γιατί αλλιώ δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ. Επίση, δεν πρέπει να αφήσουμε ε, θέματα όπω η μετανάστευση να γίνουν υπερξιακά ερωτήματα τα οποία λύνουμε μόνο βραχυπρόθεσμα. Χρειαζόμαστε καλύτερη διαχείριση των συνόρων, να προστατεύουμε αυτού που έχουν ανάγκη και να είμαστε αυστηρούς, αυστηροί με αυτού που δεν έχουν ανάγκη και ε, να είμαστε και σκληροί εναντίον αυτών που εκμεταλλεύονται του ευάλωτου. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στι αρχέ του κράτου δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών, γιατί χωρί αυτά δεν θα υπάρχει τίποτε. Δόκτωρα Φόντερ Λάιον, Καλωσορίζω τα όσα μας είπατε και να ε, είστε βέβαιοι ότι θα είμαστε εταίροι στον ευρωπαϊκό δρόμο μα. Ο κύριο ε, Λαρτουρού για ένα λεπτό. Κυρία Λάιον, ε, έχετε πολύ φιλόδοξο στόχο για την Ευρώπη να μειωθούν κατά 50% οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030. Έχετε δίκιο. Είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Για να κερδίσουμε σε αυτή τη μάχη ε, χρειαζόμαστε χρήματα. Ναι, χρειαζόμαστε μια τράπεζα για το κλίμα. Ένα σχέδιο επενδύσεων, έχετε δίκιο. Αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει να βρούμε 100 δισεκατομμύρια για το κλίμα, 100 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, για να χρηματοδοτήσουμε ένα πραγματικό σχέδιο μάσο για την Ευρώπη, ένα πραγματικό πρόγραμμα έρευνα και για να επιδοτήσουμε όλε τι οικογένειε και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Για να χρηματοδοτηθεί η μετάβαση. Πού θα βρούμε 100 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, χωρίς να υπερφορολογήσουμε τους απλούς πολίτες. Πρέπει να καταπολεμήσουμε το ευρωπαϊκό φορολογικό ντάμπινγκ. Όταν ήμουν μικρόν, ε, μικρός, οι φόροι επί των κερδών ήταν γύρω στο 40% κατά μέσο όρο. Έχει πέσει στο 20%. Ενώ τα κέρδη και τα μερίσματα εκτινάσσονται. 20% στην Ευρώπη, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες από την εποχή του Ρούσβελτ είναι στο 38%. Έχει δημιουργήσει σε τέσσερι μήνε μόνο ένα ομοσπονδιακό φόρο Ρούσβελτ. Αν θέλουμε λοιπόν να κερδίσουμε τη μάχη του κλίματο, το ερώτημα είναι, θα μπορούσαμε στα πλαίσια του προσεχού ΠΔΕΛΤΑΠΗ να έχουμε 100 δισεκατομμύρια παραπάνω το χρόνο. Μπορούμε να ζητήσουμε και οι μέτοχοι να πληρώσουν με ένα φόρο 5% μόνο και χωρί να θίξουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, χωρί να θίξουμε του ε, τις, τις, ε, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν, αρκεί, ε, δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτή την προσπάθεια για να σώσουμε το κλίμα. Ευχαριστώ, Βάουτμανς. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, κυρία Φόντερ Λάιν. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι σήμερα κάνετε μια πολύ καλή ομιλία. Πολλοί ήμασταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Και εγώ ήμουν επιφυλακτική, αλλά άκουσα μια γυναίκα που έχει πραγματικό όραμα για την Ευρώπη, ενθουσιασμό για την Ευρώπη, που θέλει να ανανεώσει την Ευρώπη συνεργαζόμενη με το Κοινοβούλιο, που θέλει να μα δώσει το, δίκαιο, τη, συγγνώμη, το δικαίωμα νομοθετική πρωτοβουλία. Βεβαίω είναι σημαντικό και που είστε γυναίκα και που είπατε ότι θα υπάρχει ισότητα ανδρών γυναικών στη Νέα Επιτροπή και θέλετε να παλέψετε κατά της ε, βίας φύλου. Κοιτάξτε, όλοι βλέπουμε πολλούς άνδρες με κουστούμια, αλλά πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε και γυναίκες ε, στα όργανα ε, λήψη αποφάσεων, αλλά η πολιτική μετανάστευση δεν ξέρω αν μας πείθει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμυνα. Ε, και αυτά που είπατε, τον Ευρωπαϊκό Στρατό, ίσως πρέπει να τα δούμε μεταγενέστερα. Κυρία Φόντερ Λάιν, ελπίζω ότι θα μπορέσετε να κρατήσετε στιβαρά τα ενία για να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα προβλήματα και για να είμαστε ισχυροί. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μουρεσάν, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε υποψήφια, πολλά υπόθηκαν. Θα ασχοληθώ με τα εξή. Πρώτον, να σας συγχαρώ. Διότι επιτύχατε τη σωστή ισορροπία για την ενεργειακή πολιτική, την κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα στον τομέα αυτό. Πρέπει να βελτιώσουμε την ενεργειακή μας απόδοση, να μειώσουμε τις εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα και όλα αυτά πρέπει να γίνουν με υπεύθυνο τρόπο Έχοντα υπόψη το οικονομικό, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των μέτρων μας και ε, ε, ιστάμενοι ε, στο πλευρό των λαών, στο πλευρό των περιφερειών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Προτείνεται ένα φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό πρόγραμμα. Σωστό είναι νομίζω και το στηρίζω. Επίση, προτείνεται ένα ε, ε, μέσο σύγκλησης για την Ευρωζώνη. Αλλά σας παρακαλώ το μέσο αυτό να είναι ανοιχτό και για χώρε που δεν είναι ακόμη στην Ευρωζώνη, αλλά που προετοιμάζονται να ενταχθούν, για να επιτρέψετε σε αυτέ τι χώρε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέσου αυτού, να αποφεληθούν από τη λειτουργία του και να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων. Θα του επιτρέψει την ένταξη στην Ευρωζώνη. Θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή οικονομία κάτι τέτοιο και επίση θα βελτιώσει την ενότητα παντού στην Ένωση. Και τρίτον, ω ε, Μια λέξη Σέγγεν. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούν τις συνθήκες ε, ένταξη στο Σέγγεν από το 2011 και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε επανειλημμένα ζητήσει να ενταχθούν. Σας παρακαλώ να είστε στο πλευρό του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και μαζί να αξιοποιήσετε τι δυνατότητε που έχετε στη διάθεσή σα, ούτω ώστε η Βουλγαρία και η Ρουμανία να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν. Είναι το ένα θέμα που οι πολίτε αυτών των δύο χωρών αναμένουν κυρίω από την Ένωση. Θα βελτιώσει την ασφάλεια του χώρου Σέγγεν, δεν θα την αποδυναμώσει. Και, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε ένα κοινοβούλιο με πολύ διαφορετικές απόψεις. Αλλά από ό,τι είδα σήμερα από την κυρία υποψήφια, από αυτά που είπε, έλαβε όλες μας τις θέσεις υπόψη και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει να τη στηρίξει το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ζωχίνιο. Κάρλος, ένα λεπτό. Κυρία Φοντελάιεν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί απευθείας ε, τους ε, Ευρωπαίους πολίτες και ως ε, Πορτογάλος σοσιαλιστής εκπροσωπώ ψηφοφόρους που επιθυμούν ένα προοδευτικό πρόγραμμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στην ομάδα μου είχα σοβαρές επιβολίες για το κατά πόσο το επίπεδο δέσμευσής σας είναι εφάμιλο με, αυτό τις δεσμεύσεις που εμείς η Πορτογαλική Αντιπροσωπεία έλαβε απέναντι στους ψηφοφόρους της. Ε, βέβαια, από τις γραπτές σας απαντήσεις και από τη σημερινή σας ε, ομιλία επίστηκα αρκετά περισσότερα, ήταν πολύ πιο πιστικά. και γι' αυτό είμαστε σε, σε, στην κατάσταση να περάσουμε προς ένα άλλο, ένα άλλο επίπεδο, σε, ένα σε μια άλλη φάση, τη φάση της ε, συγκεκριμενοποίησης. Γι' αυτό και θα θέλαμε ένα φιλόδοξο πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο που θα προωθεί τη σύγκληση και την ε, συνένεση με ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη. Τι θα κάνετε για κάτι τέτοιο, πώ θα δώσετε κίνητρα για τη μεταρρύθμιση τη Ευρωζώνη και για τη δημιουργία ενό ε, ε, εύρου του προπολογισμού ώστε να προστατεύσει την Ευρώπη από συστημικές κρίσει. Πώ θα μετατρέψετε τι θετικέ δεσμεύσει που αναλάβατε σε συγκεκριμένε πολιτικέ για να επανασυνδέσουμε του ευρωπαίου πολίτε με αυτό το καταπληκτικό Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό σχέδιο. Κυρία Φοντερ είναι ώρα για δράση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ιντφελτ, Σοφία, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φοντερ Λάιεν, ε, είμαι απόλυτα πεπισμένη για τα προσόντα σας. Εδώ, εδώ στη μέση βρίσκομαι. Είμαι η κόκκινη βούλα στη μέση του ημικυκλίου πιστεύω ακράδαντα τα προσόντα και την αξία σας. Το θέμα είναι, όχι αν είστε το σωστό πρόσωπο, αλλά το σωστό πρόσωπο για τη συγκεκριμένη θέση. Και εκεί δεν έχω πιστεί ακόμη απόλυτα. Η πρότασή σα καταρχήν για μηχανισμό κράτου δικαίου. Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση αυτή είναι ανεπαρκή, αδύναμη, με υπερβολικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογή. Και Κανονικά ο κύριος μας ε, θα το πρότεινε κάτι τέτοιο και ε, είχα ε, μια ευκαιρία να το εξετάσω. Επίση, πώ θα καταπολεμήσετε το ρατσισμό και την ξενοφοβία που είναι μείζον πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Και τρίτον, δεν με προβληματίζει τόσο το θέμα των σωστών πολιτικών, γιατί συμφωνώ με τις προτάσεις σας. Η εφαρμογή όμως, η συγκεκριμενοποίηση των πολιτικών είναι το πρόβλημα, γιατί είμαστε πολύ ικανοί στην εκπόνηση κανόνων, αλλά δύσκολοι στην εφαρμογή. Dieselgate, ε, σκάνδαλα προστασίας δεδομένων από το Facebook, ε, νομοποίηση όδων από παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις ε, κράτους δικαίου στην Ουγγαρία, Πολωνία και αλλού. Οι προηγούμενες ε, Ευρωπαϊκές Επιτροπές, ε, οι προηγούμενοι μάλλον, ήταν αρκετά άτολμοι. Και φαίνεται ότι λόγω της διαδικασία που ακολουθήθηκε είσαι περισσότερο εκπρόσωπος των κρατών μελών. Όπως ε, προηγούμενοι Επίτροποι, θα είστε απλώς το φερέφωνο αυτών των κρατών μελών ή μάλλον ένα ε, πυθύνιο πλάσμα ή θα γίνετε πραγματικά αυστηρίο που θα θέλαμε να είστε στα ευρωπαϊκά θέματα. Κυρία Τσάντερ, κυρία υποψήφια, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα ε, είναι ιστορική στιγμή, διότι θέτουμε τις κατευθύνσεις για τις, ε, την επόμενη πενταετία και είναι ταραγμένη περίοδος. Οι συμμετοχή σε εκλογές αποδεικνύουν ότι οι συμπολίτες μας ε, ενδιαφέρονται εκ νέου περισσότερο για την Ένωση, αλλά αναμένουν από εμά λύσεις, εγγυήσεις για την ευημερία τους, την ελευθερία και την ασφάλειά τους. Μια Ευρώπη που τους προστατεύει, όπως ε, ήταν και το έμβλημα της Αυστριακής Προεδρίας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η ισχυρότερη πολιτική δύναμη και θέλουμε να διαμορφώσουμε ακριβώς τη διαδικασία αυτή. Και τη διαδικασία βεβαίως ε, ορισμού υποψηφίου που βεβαίως είναι επικρίσιμη και αυτό έχει οδηγήσει σε απώλεια εμπιστοσύνη. Αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε τη διαδικασία από το άτομο που προτείνεται τώρα. Το θέμα είναι γρήγορα να επανέλθει αυτή η εμπιστοσύνη των ε, συμπολιτών μα. Πρέπει να βλέπουμε προ τα μπρό. Πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό χρειάζεται για να καταργήσουμε τι καθυστερήσει, να υπερβούμε τι καθυστερήσει. Και ε, χαίρομαι που θέλετε να υπάρξει νομική βάση για το σύστημα speech and candidate στο μέλλον, γιατί οι πολίτε θα πρέπει να το δεχτούν, να το στηρίξουν. Πρέπει να του δείξουμε ότι οι αποφάσει που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι διαφανεί. Χρειαζόμαστε ένα όραμα για την Ευρώπη. Αλλά και προσωπικότητε, που να είναι διατεθειμένες να αναλάβουν τις ευθύνες αυτές. Να δράσουν ενεργά για να διαμορφώσουν το μέλλον, να εφαρμόσουν όσα αποφασίζουμε. Με εσά έχουμε ένα άτομο που ως επικεφαλής της Κομισιόν θα είχε δυνατότητα να επιβάλλει την πολιτική σα. Και όχι μόνο μα πείσατε σήμερα γι' αυτό. Κάποιοι είμαστε πεπισμένοι, αλλά κάποιοι πιστήκαν και σήμερα. Γι' αυτό θα έχετε την πλήρη υποστήριξή μας. Και νομίζω ότι προτείνετε τα σωστά θέματα, εστιάζετε σωστά επιθεμάτων που δεν είχαν ε, ε, αποτελέσει προτεραιότητα μέχρι τώρα, όπως για παράδειγμα η βία κατά των γυναικών. Θα σας στηρίξουμε πλήρως. Ευχαριστώ πολύ. Σίντερ, ένα λεπτό. Σας παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φόντελάιν, ε, ήμουν ιδιαίτερα επικριτικός έναντι της διαδικασίας ε, μέσω της οποίας ε, προταθήκατε, αλλά παρόλα αυτά η ομιλία σας είχε πολλά σωστά σημεία. Αλλά με το χέρι στην καρδιά πρέπει να πω ότι έχουμε ακούσει πολλούς καλούς λόγους στην Ευρώπη. Το σημαντικό είναι συγκεκριμένα εγχειρήματα. Για παράδειγμα, να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη, η φοροαποφυγή, νόμιμη ή παράνομη πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να ληφθούν ουσιώδη μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει επιτέλου ο κοινωνικό πυλώνα να γίνει πραγματικότητα στην Ευρώπη. Και εδώ είναι το θέμα. Ακριβώ η εφαρμογή πολύ συχνά αποτυγχάνει. Και κυρίω αποτυγχάνει λόγω κάποιων κρατών μελών. Γιατί τα μισά έχουν συντηρητικέ κυβερνήσει δηλαδή οι κυβερνήσει ε, των κομμάτων που συμμετέχουν στο ΕΛΚ. Οπότε αυτή η εφαρμογή που είναι το αποφασιστικό μας ε, απασχολεί. Και τελευταίο, αλλά όχι και ασήμαντο, για το κράτος δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο να μιλάμε, αλλά να διασφαλίζουμε και εσείς θα πρέπει ως πρόεδρο τη Επιτροπή να διασφαλίσετε ότι στην Ευρώπη δεν θα υποχωρεί στο μέλλον έναντι των ε, Όρμπαν και των Σαλβίνη. Ευχαριστώ, Γκέρενς. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φόντερ Λάιν, όταν βλέπω τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πραγματικά απογοητεύομαι. Όταν βλέπω όμως τις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρηγορούμε από τότε που ο Μπάρακ Ομπάμα δεν είναι πλέον πρόεδρος ε, ε, έχουμε χάσει την κατεύθυνσή μας ε, και η πολυμορφία πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν μια θέση που χειρεύει. Ποιος θα την αναλάβει. Η Ευρώπη θα το κάνει αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις υπεύθυνε δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το χάσμα που υπάρχει βορρά-νότου και αναλωτικής δύσης. Επίσης, ξεκινώντας από τις ε, παγκόσμιες προκλήσεις, ε, για παράδειγμα το κλίμα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την Κίνα, την Ινδία και τη Μέση Ανατολή, αλλιώς ε, μια οικονομία χωρίς άνθρακα θα αποτελέσει απλώς ουτοπία. Θα πρέπει να τολμήσουμε. Εάν εκλεγείτε και αν τα καταφέρετε, το οποίο σας το εύχομαι, κανείς στο τέλος της θητείας σας δεν θα σας ευχαριστήσει. Εάν όμως ε, τελικά αποτύχεται, κάτι το οποίο απέφχομαι, εμείς ε, θα μας κατηγορούν όλους, θα μας στείλουν στο διάολο πραγματικά. Και επομένω ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Μάινταλ για 1,5 λεπτό. Κυρία υποψήφια για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε η Ευρώπη να φτάνει στον κάθε Ευρωπαίο. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο Βρυξέλλες ή Στρασβούργο. Ευρώπη είμαστε όλοι μας. Η Ευρώπη λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι περισσότερη για μερικούς και λιγότερη για άλλους. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η Ευρώπη να φτάνει σε κάθε χωριό, πόλη, σε κάθε αγόρι και κορίτσι, σε κάθε πολίτη, ε, σε όλους τους πολίτες χάρη σε συγκροτημένο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και πρωτοβουλίες. Κανένας Ευρωπαίος δεν θα πρέπει να εγκαταλείπει την πατρίδα του, την περιοχή του για οικονομικούς λόγους. Και οι κανόνες να ισχύουν για όλους. Και όταν χώρες όπως η Βουλγαρία πληρούν τα κριτήρια του Σέγγεν, θα πρέπει όντως να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν. Θα έχετε λοιπόν συνομιλίες με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, με κράτη-μέλη που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν ότι η Βουλγαρία έχει πληρώσει τα κριτήρια για την Ευρωζώνη, για να μην θεωρηθεί μια κλειστή λέσχη. Ε, πιστεύετε ότι όταν οι χώρες πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να διευρυνθεί η Ευρωζώνη την επόμενη πενταετία. Επίσης, ε, ε, κάθε επιχείρηση, κάθε επιχειρηματίας, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση έχει πρόβλημα να βρει καταρτισμένους και επιδέξιους επαγγελματίες. Δεν θα πρέπει να είμαστε λοιπόν λίγο πιο φιλόδοξοι και να θετήσουμε αποφασιστικές δράσεις για να αναβαθμίσουμε τα επαγγελματικά προσόντα των συμπολιτών μας. Μετά τη σημερινή μέρα θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ σημαντικό να περάσουμε από τα λόγια στα έργα και θα συμπορευθώ μαζί σας ώστε να έχουμε μια σταθερή ενεργειακή αγορά, μια μελλοντοστραφή και ε, εξυγχρονισμένη ε, βιομηχανία, μια ε, βιομηχανία που θα σπάζεται τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, ώστε να εξασφαλίσουμε ακόμη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα για την ήπειρό μας. Ευχαριστώ κυρία Σχάλντε για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ομιλία σας κυρία Φόντερ Λάιεν και σας ευχαριστώ που τίνατε βίκονου στα αιτήματα των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Την, περιβαλλον... την κλιματική πολιτική, μείωση ε, των εκπομπών διοξίδιων του άνθρακα μέχρι το 2030. Για να ελοπίσουμε όμω του στόχου μα, θα πρέπει να φροντίσουμε να δράσουν και τα κράτη-μέλη. Στι σκανδιναβικέ χώρε έχουμε τρει σοσιαλδημοκρατικέ κυβερνήσει. Εμεί θα προωθήσουμε αυτά τα μέτρα. Στη Δανία έχουμε νέα κυβέρνηση και μιλούμε για 70% μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030. Οπότε πρωτοστατούμε. Ελπίζω να περάσουμε στις δράσεις και στα έργα, να απαγορεύσουμε τα διζελοκίνητα οχήματα. Ε, θα πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα να είμαστε αποτελεσματικοί και φιλόδοξοι στις πολιτικές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ω μια κοινότητα άνθρακα και χάλιβα. Ελπίζουμε, κυρία Φοντερ Λάιεν, να πρωτοστατήσετε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα γίνει μια Ευρωπαϊκή Ένωση του κλίματο και θα βρεθούμε στο πλευρό σα γι' αυτό. Η κυρία Γκάμον για ένα λεπτό. Um, κυρία Φοντερ Λάιεν, ελπίζω πραγματικά να επιτύχετε. Δεν είναι πεπισμένη ε, σήμερα, αλλά ελπίζω να πιστώ μέχρι το τέλο τη θητεία. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, να καθορίσουμε την ψηφιακή εποχή μέσω ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Δεν πρέπει να απογοητεύουμε τους ανθρώπους ε, περιοριζόμενοι στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή να τους εκπλήξουμε με τη φιλοδοξία μας στηρίζοντας ε, πολύ ευρύτερους στόχους, τον πιο φιλόδοξο στόχο που μπορούμε να καθορίσουμε από κοινού. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που θέσατε, αλλά το κύριο εμπόδιο δεν είναι εδώ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά κυρίως το Συμβούλιο. Και το Συμβούλιο είναι το θεσμικό όργανο που ενισχύθηκε μέσω όλης αυτής της διαδικασίας ορισμού του Πρόεδρου της Επιτροπής και λυπάμαι που αποφεύγουμε τις συζητήσεις για κάποια θέματα. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θίξουμε ακριβώς τα σημεία που πονάνε. Γιατί αυτά πρέπει να αλλάξουμε. Διότι το Μάιο η ψήφος ήταν ψήφος ανανέωσης μεταρρύθμιση τη Ένωση, να λειτουργεί καλύτερα. Πραγματικά πρέπει να λειτουργεί καλύτερα για τους ε, πολίτες ε, της. Πρέπει λοιπόν να μεταρρυθμίσουμε και να ανανεώσουμε την Ένωση, γιατί αλλιώς όλα τα οράματα που μας παρουσιάσατε δεν θα ε, υλοποιηθούν. Ευχαριστώ. Κύριος Κόρμπετ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα σχόλια για τη δημοκρατία που έγινε από τα άδεια έδρυνα τώρα ε, πίσω στο ημικύκλιο με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εσείς κυρία Φόντερ θα αναλάβετε καθήκοντα μόνο εάν σας εγκρίνει η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενώ την επόμενη εβδομάδα στη Βρετανία θα αναλάβει ένας Πρωθυπουργό ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να υπάρξει κάποια θετική ψήφος υπέρ του στο Κοινοβούλιο ε, στην Αγγλία. Και αυτό πραγματικά είναι μία αντίθεση που μας σοκάρει όλους ε, εσείς ε, ε, αν αναλάβετε καθήκοντα θα υποχρεώσετε την το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαναχωρήσει σε μια αρχή που είχε υποστηρίξει το Spitzer Candidate και επομένω ε, θα πρέπει να κάνετε πολλά από αυτά τα οποία ζητά το Κοινοβούλιο και αυτά τα οποία είπατε για την πολιτική είναι σημαντικά, το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι επίσης σημαντικό και επίσης να πω και ότι είπατε για τον Brexit είναι σημαντικό. Ότι δέχεστε την ανάγκη να υπάρχει παράταση στην προθεσμία για ε, εύλογου. Ε, εύλογε αιτίε. Και να σα πω ότι υπάρχει σωστή αιτία. Το βρετανικό κοινό αλλάζει γνώμη για το Brexit. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που εξελέγησαν ε, πρόσφατα έχουν ε, άλλη άποψη. Οι δημοσκοπήσεις επίση δείχνουν ότι αλλάζουν τα πράγματα. Όλοι όσοι βρίσκονται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ζητούν νέο δημοψήφισμα και πραγματικά αφήστε ανοιχτή αυτή την πόρτα, αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Ο Πέδρο Μάρκες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φοντερ η δέσμευσή σας ε, και προφορική και γραπτή για περισσότερη ανταγωνιστικότητα, για μια βιώσιμη και αλληλέγγυα Ευρώπη, δείχνει ότι μπορέσετε να διαβλέψετε σωστά το πρόγραμμά μας και μπορέσετε να διαβλέψετε και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων. Η Ευρώπη χρειάζεται κατεπίγουσα δράση και επομένως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν διστάσατε να αναλάβετε δεσμεύσει, οι οποίες οδεύουν προς την κατεύθυνση που περιμένουν οι πολίτες. Σαφείς δεσμεύσεις, σαφή επιτεύγματα. Ε, ελπίζουμε όμω ότι θα έχετε και τη δυνατότητα να συμβιβαστείτε και να αποφύγετε ε, το ε, μπλόκο που επιβάλλουν αρκετές χώρες ε, του Συμβουλίου. Για την Ευρωζώνη, για το περιβάλλον δεν υπάρχει περιθώριο για δισταγμού. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές όπως για παράδειγμα την έγκριση ενό κατάλληλου προπολογισμού για την Ευρώπη. Ε, θεωρούμε ότι τα όσα είπατε σήμερα και όσα μας γράψατε αποτελούν μεγάλες προσδοκίες ε, και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει και ό,τι μπορεί από πλευρά του. Οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιμένουν τίποτα λιγότερο από εμά. Επομένω, η δέσμευσή σα σήμερα ε, είναι οριστική. Οι Ευρωπαίοι ζητούν πέντε χρόνια ε, εξηλαίωσης του ευρωπαϊκού οράματος μετά από 10 χρόνια κρίσης και δισταγμών. Ας ε, ε, επανικοδομήσουμε από εδώ και πέρα την Ευρώπη των ονείρων μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση και τώρα θα έχουμε την απάντηση της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Mr. President, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τόσο ζωηρή συζήτηση ήταν επικοδομητική, εκφράστηκαν διαφορετικές απόψει και αν χρειαζόταν απόδειξη ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη είναι ολοζώντανη, εσείς μας τη δώσατε σήμερα εδώ στο σώμα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Επανελειμμένα αναφέρθηκε ότι μόνο δύο εβδομάδες είχαμε για να γνωριστούμε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που είχα αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα μου. Βεβαίως ε, ε, μια ομιλία είναι μόνο μια ομιλία. Αλλά νομίζω ότι λάβατε σήμερα και τις καθευτήριες γραμμές, ε, τις γραπτές αναλυτικές καθευτήριες γραμμές για τα θέματα για μια κλιματικά ουδέτερη την Ευρώπη το 2050, μια πιο κοινωνική και ανταγωνιστική Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της, μια Ευρώπη που θα δώσει νέα όθηση στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, μια ισχυρή Ευρώπη που υπερασπίζεται τον ευρωπαϊκό μας τρόπο ζωή. Ακούγοντα σας, άκουσα πολλά επιχειρήματα και έχω πλήρη συνέστηση ότι έχουμε αυτή την αίσθηση ότι υπάρχουν ε, διαφοροποίησεις μεταξύ Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Πρέπει να υπερβούμε αυτές τις ε, διαφοροποίησεις. Έχω κάθε σεβασμό γιατί γνωρίζω τις προσπάθειες που έγιναν στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και που συνεχίζουν να κάνουν για να ενταχθούν στην Ένωσή μας, στο Σέγγεν, στην Ευρωζώνη και νομίζω ότι όταν πληρούνται τα κριτήρια πρέπει να ανταμείβονται. Επίσης, γνωρίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ε, χάσματα σε έναν βαθμό μεταξύ βορρά και νότου και έχω εξηγήσει πώς θα μπορούσαμε να τα υπερβούμε, πώς θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ε, υπευθυνότητας και ε, ευελιξίας, ε, ούτως ώστε να επιτύχουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη που χρειαζόμαστε. Θέλω να έχω πολύ πιο στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό στηρίζω το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε υγιείς τρόπους ούτως ώστε να εδραιωθεί το σύστημα Spitzenkandidat. Είμαι πεπισμένο ότι μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω να υπάρξει ανανεωμένη εμπιστοσύνη, συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Είμαι ο φυσικός ασύμμαχος σύμμαχος, ε, ας το πω έτσι. Και, σε τελευταία ανάλυση, πριν ψηφίσετε σήμερα, να καταλήξω με μια δήλωση πάλι ενός Έλληνα, Έλληνα μεγάλου πολιτικού που είναι ένας ε, από τους ιδρυτές της δημοκρατίας. Είναι μια θαυμάσια δήλωση για την κοινή μας εργασία. Λέει το μυστικό για την ευημερία και το μυστικό για την ελευθερία είναι το θάρρος. Ελεύθερον μεν, εύδεμον μεν το ελεύθερον, ελεύθερον δε το εύψυχον. Αυτό πρέπει να είναι και το έβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Φόντερ Λάιεν. Πέρα τη συζήτηση, ε, γνωρίζετε ότι η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 6 το απόγευμα. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3. Ευχαριστώ πολύ.